Guten Tag. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Αγαπητοί συνάδελφοι, τα πρακτικά τη συνεδρία χθε και τα κείμενα είναι διαθέσιμα, υπάρχουν παρατηρήσει, δεν βλέπω κανέναν να ζητάει το λόγο. Εγκρίνω λοιπόν τα πρακτικά αυτά τη συνεδρίασης. Δύο ομάδες, και η